colleagues, an excellent good afternoon. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Uh, not only a little bit, but really fit for everything that is coming up right now. So I'm... Ελπίζω να είστε έτοιμοι και σε φόρμα για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας σήμερα. Και φυσικά όσοι συμμετέχετε στη συνεδρίαση από το σπίτι, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 6 παρατέταρτο. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εδώ έχω να προτείνω μία αλλαγή, να αλλάξουμε κάπως τα σημεία και να εξετάσουμε πρώτα το σημείο 5, Γενικό Προϋπολογισμό, και έπειτα το σημείο 4 την πολιτική συνοχή. Δηλαδή 1, 2, 3, 5, 4. Εάν ε, συμφωνείτε όλοι μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ανακοινώσεις της Προέδρου οι οποίες είναι σύντομες. Θα ήθελα όμως να πω τα εξή. Ζούμε σε μια ιδιαίτερα συνήθιστη εποχή όλοι μας ε, το ζούμε στις χώρες μας και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο στον ε, τομέα της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Βέβαια, η κατάσταση ε, διαφέρει. Στη δική μας επιτροπή το κύριο θέμα είναι τα δικαιώματα των γυναικών ισότητα των φίλων και βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση. Η επιτροπή μας επομένως θα πρέπει να ακούγεται και να έχει μέλη ενεργά. Αυτές λοιπόν είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ που έχω να σα δώσω για τους επόμενους μήνες. Κοιτάζουμε λίγο τα θέματα. Έχουμε την βία κατά των γυναικών, όπου έχουμε το παράδειγμα αυτών των θαραλέων γυναικών στη Λευκορωσία, που μας ε, λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για την παρουσία μας ε, και την παρουσία σας στις συνεδριάσεις ε, που κάνατε ό,τι μπορούσατε έτσι ώστε να είμαστε λειτουργικοί. Επίσης, μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας. Από τώρα δηλαδή, από 5 παρα 6 μέχρι τις 7 όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή, είτε εδώ στην αίθουσα είτε εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας τους ε, καταλόγους ψηφοφορίας που θα έχουν εκτυπώσει. Περνάμε τώρα στο σημείο 3, την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Έχουμε 80 τροπολογίες, αρκετή δουλειά έχει γίνει δηλαδή. Η συγγήτρια πρότεινε 12 συμβαστικέ τροπολογίε. Η συντάκτρια της νομοδότηση είναι η Μαρία Νταγκράσα Καρβάλιο και επί τη ουσία ε, η συγγήτρια η Σαμπίνα Φερχάιν από την Επιτροπή Πολιτισμού. Γνωρίζετε την διαδικασία, πρέπει να την έχετε συνηθίσει τώρα. Έχετε λάβει τους κατάλογους ψηφοφορίας και τις οδηγίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε αν υπάρχει απαρτία. Όσοι είστε στην αίθουσα σηκώστε το χέρι, όσοι συμμετέχετε εξ αποστάσεως πιέστε το ανάλογο κουμπί. Τώρα σας παρακαλώ για να δούμε εάν υπάρχει απαρτία. Η γραμματεία με ενημερώνει ότι υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ξεκινά η ψηφοφορία, επομένως, στις 5, όπως είπα, μέχρι τις 7. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως ε, κάνουμε τελευταία. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει την πέμπτη. Δεν είναι ακόμα πέντε, οπότε θα ξεκινήσουμε σε τέσσερα λεπτά. Από τις πέντε μέχρι τις εφτά οι ψηφοφορίες λοιπόν. Και όλα θα γίνουν όπως σας ανέφερα. Και με αυτό περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το σημείο 5, Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, όλα τα τμήματα. Η συγητής της εγγνωμοδότησης είναι ο Ρομπέρτ Μπιεντρόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ στην αίθουσα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 9η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα δώσω όμως ευθύ αμέσω το λόγο στον Ρόμπερτ και έπειτα στους σκιώδεις εισηγητέ εφόσον το ζητήσουν. Ρόμπερτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Ευελέν, χαίρομαι που σας βλέπω όλους ε, για το θέμα των γυναικών στη Λευκορωσία που το αναφέρατε. Ως Επιτροπή πρέπει να εκφραστούμε κάπως υπέρ τους. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή χρειάζονται την υποστήριξή μας, γιατί είναι πραγματικά φανταστικό που κι εσείς αναφερθήκατε σε αυτό και το θυμήσατε. Τώρα, για το χρήμα. Τον Ιούλιο εγκρίναμε μια σειρά από τροπολογίες από του προπολογισμού για τον προπολογισμό το 2021. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους μου τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Όλες κέρυες και είχαμε και πολύ αποτελεσματική συνεργασία. Ε, ανέλαβα την εντολή να επιφέρω κάποιες απαραίτητες ε, προσαρμογές βελτιώσεις στην πρόταση βάσει της θέσης του Συμβουλίου που προέκυψε το καλοκαίρι. Όσο για τη γνωμοδότηση που συζητούμε σήμερα αφορά το ψήφισμα που θα συνοδεύει το Γενικό Προπολογισμό για το 2021 και αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που υποβλήθησαν στην Επιτροπή μας. Το βασικά θέματα που θίγει η έκθεση είναι πρώτον ότι είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας ε, η ευθυγράμμιση της διάστασης του φύλου και η συμπερίληψη της διάστασης του φύλου όπου συζητάμε για χρήμα, κονδύλια και ούτω καθεξής, πρέπει να υπάρχει αυτή η διάσταση, το mainstreaming για τα δύο φύλλα. Ε, έπειτα, για τα θέματα που ανέφερες, αναφέρατε Εύελιν, χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να καταπολεμήσουμε την έμφυλη βία, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19. Βλέπουμε να διωγγώνονται τα φαινόμενα βίας κατά των γυναικών και παιδιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πρότασής μας. Επίσης, πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Ταμείου ΣΥΝ, ιδίως και στο πλαίσιο του COVID-19. διότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα και όποτε βλέπουμε ένα κύμα ε, γεγονότων που, που είναι, απόρρια κάποιες κρίσεις, οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα συνήθως και πολύ συχνά αυτό παραβλέπεται. Επίσης προτείνεται η άξια του προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Ισότητας των Φύλων με περισσότερες δεσμεύσεις για πληρωμές και για τις ε, οργανώσεις των δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι λοιπόν σημαντικές όλες αυτές τις τροπολογίες ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, όπως ανέφερε και η κυρία Τερ, είναι ε, η προθεσμία στις 9 Σεπτεμβρίου, την 5η στις 12 την Τετάρτη, συγγνώμη, στι 12. Ε, λόγω του περιορισμένου χρόνου, δυστυχώ οι τροπολογίε μπορούν να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Η ψηφοφορία προβλέπεται 21-22 Σεπτεμβρίου και σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι βάσει των ε, κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Προπολογισμού οι τροπολογίες θα πρέπει να ε, έχουν να κάνουν ε, με τα θέματα των τροπολογιών που προέκυψαν τον Ιούλιο Αυτά από μένα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω αμέσω το λόγο στους σκιώδει εισηγητές, την σκιώδη του ΕΛΚ, την κυρία Πίτικανεν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Α, δεν είναι συνδεδεμένη κυρία Πιτικάινεν. Πρέπει να πω ότι στην οθόνη βλέπω τα ονόματα από εδώ μακριά, αλλά όχι τόσο μακριά, διότι δεν έχω και την απαραίτητη ικανότητα στην όραση. Η κυρία Πιτικάινεν δεν είναι συνδεδεμένη, οπότε θα πρέπει να περάσουμε στον επόμενο στον κατάλογο των ομιλητών. Ραφαέλα, η κυρία Ραφαέλα για του Ρινιού. Διότι μόλις διάβασα ότι η κυρία Τολρέ δεν θα είναι εδώ. Γεια σας, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θα μιλήσω εκ μέρους της Ιρέν. Η κυρία Τολρέ είναι η σκιώδης εισηγήτρια από την πλευρά των, ε, της ομάδας Renew. Η γνωμοδότηση αυτή εξετάζει τις τροπολογίες από τον από τον Ιούλιο πολλά από τα σχόλια μας έχουν ληφθεί υπόψη όπως καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και η καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης της πανδημίας του COVID. Επίσης, βελτιωμένη ε, πρόσβαση στα κονδύλια ε, για την ευθυγράμμιση της διάστασης του φύλου και από τους ε, ΛΟΑΚ και Κάτι που είναι σημαντικό για μας στη γνωμοδότηση είναι η προφορική παρουσίαση για τα θέματα των γυναικών στην, στον κλάδο των ICT. Η προφορική αυτή παρουσίαση θα επηρεάσει τη συμμετοχή τους ε, και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά κυρίως τη διάσταση της ψηφιοποίηση. Επίσης πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παράγραφο για τα δικαιώματα ε, της ε, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να λάβουμε υπόψη ότι όχι μόνο το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που αναφέρεται ε, στο, στην γνωμοδότηση, αλλά και το Ίδρυμα για τα Θεμελίδια Δικαιώματα κάνει πολύ καλή δουλειά για τις μειονότητες, την προστασία τους και τους ΛΟΑΚ κυρίω. Για τις τροπολογίες λοιπόν αυτές επί του, επί του προπολογισμού ζητούμε να είμαστε υπέρ των περισσότερων και ζητούμε και αύξηση του προπολογισμού του, Ινστιτού, του Ιδρύματος για τα Θεμελίδια Δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Επόμενη στον κατάλογό μου, κυρία Άντερσον από την ομάδα ID. Μόλις ενημερώνομαι ότι δεν είναι συνδεδεμένη, οπότε να δώσω το λόγο στην κυρία Βάνα από τους Πρασίνους. Ούτε εκείνη είναι συνδεδεμένη. Από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, η κυρία Γιαντβίγκα Βυσνιεύσκα. Είστε συνδεδεμένοι. Ούτε εσείς είστε συνδεδεμένοι. Οπότε προχωρούμε γοργά. Αλλά μπροστά μου βλέπω, και γι' αυτό θα έχω τη, χαλα... τη χαρά να της δώσω το λόγο, την κυρία Περέιρα από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά του και να ξεκινήσω από το γεγονός ότι είναι κρίμα που δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες στη δική μας τη γλώσσα. Η πολυγλωσία απειλείται και θα ήταν επιθυμητό να μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες στη μετρική μας γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για την πραγματική καταπολέμηση της αύξησης του αριθμού γυναικών που πέφτουν σε συνθήκε ένδυα, για την υποστήριξη των πολιτικών σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για τα σχετικά δικαιώματα των γυναικών που πρέπει να ενισχυθούν, το ανέφερε ο εισηγητή ήδη, καταπολέμηση όλων των μορφών βία κατά των γυναικών και παιδιών, καταπολέμηση τη εμπορία επίση των ανθρώπων, που συνήθω έχει θύματα γυναίκε και νερά κορίτσια, που είναι θύματα σεξουαλική εκμετάλλευση Επίση, θέλουμε να ενισχυθεί ο προπολογισμό ε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλει κανείς άλλο το λόγο παρακαλώ τώρα. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο, ούτε στην αίθουσα, ούτε εξ αποστάσεως. Οπότε, θέλω και εγώ να πω δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρεμβάσεις οι τροπολογίες ε, φαίνεται ότι συνάδουν με τόσα αναφέρονται και στο κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι όσοι κινδυνεύουν δεν πρέπει να ξεχαστούν, αλλά αντίθετα να έχουν την πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν το έργο μας πρέπει να είναι και να στηρίξουμε τη γνωμοδότησή μας αυτή, αλλά και να φροντίσουμε να ενημερώσουμε και άλλες επιτροπές για τις τροπολογίες μας ώστε να τις στηρίξουν. Ένα θέμα θα αναφέρω εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που κάνει εκπληκτική δουλειά. Μας δίνει δεδομένα τα οποία τα χρειαζόμαστε για το πολιτικό μας έργο. Πρέπει να έχουν όμως και κατάλληλη χρηματοδότηση. Και αν συγκρίνουμε υπάρχουν τόσα πολλά Ινστιτούτα και οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το συγκεκριμένο Ινστιτούτο μας ανοίγει τα μάτια και μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας δίνει. Γι' αυτό αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ σωστό και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ρόμπερτ, μήπως θέλεις και πάλι το λόγο για να προσθέσεις κάτι. Όχι, Ρόμπερτ, όλα έχουν υποθεί. Ωραία. Καλώς τότε να πούμε πάλι ποιες είναι οι προθεσμίες για τις τροπολογίες. Το είπαμε, μάλλον, οπότε σταματάμε εδώ και περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής. Η Ρέγγι είναι η αρμόδια επί Επιτροπή με συγγήτρια την κυρία Μόνικα Βάνα και η δικιά μας συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Λένα Ντυπον. Οπότε της δίνω και το λόγο. Ευθύ αμέσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρωτού αναφερθώ στην γραμμοδότηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Γραμματεία για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά το στάδιο της ε, συζήτησης σχετικά με την προετοιμασία της γραμμοδότησης. Σε γενικές ε, γραμμές έχω να σας πω ότι έχουμε χωρίσει ε, σε δύο μέρη την γραμμοδότηση, σε ένα γενικότερο και σε ένα που αναφέρεται στον κορονοϊό. προσπαθούμε να αναλύσουμε το θέμα της ε, ισότητας σε όλους τους κύκλους πολιτικής ε, και στους ε, διαγωνισμούς. Επισημαίνουμε ότι χρειάζεται αναθεώρηση και επανεξέταση ορισμένων πτυχών των δημόσιων διαγωνισμών και το ίδιο ισχύει για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη. Στην Επιτροπή Συνοχής πρέπει να προσέχουμε να υπάρχει ίση εκπροσώπηση ε, των ε, φύλων, γι' αυτό μπορούμε να προτείνουμε συγκεκριμένα όργανα, θέματα κατάρτισης, ας πούμε, εκπαίδευσης, έτσι ώστε η εφαρμογή της ισότητας ε, των φύλων σε όλους τους κύκλους πολιτικής να γίνει πραγματικότητα και να μην χάσουμε ευκαιρίες. Επίσης, καλούμε και τα κράτη-μέλη με τις αρμόδιες αρχές να ενεργοποιηθούν, να προσπαθήσουν τα ίδια με διάφορες εκστατείες ευαισθητοποίησης και διάφορα σχετικά προγράμματα να περάσουν την ε, έννοια της ε, ισότητας σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό χρειάζεται τεχνογνωσία, Βέβαια, αυτό θα γίνει από τη βάση προς τα πάνω και όχι με την υφιστάμενη πρόταση top-down, από πάνω προς τα κάτω. Μετά, περνάμε στο σκέλος του κορονοϊού. Η κρίση που ήρθε από τον κορονοϊό έχει αλλάξει πάρα πολλά στις ε, ζωές μας. Εδώ η πολιτική συνοχής ε, οφείλει και ε, θα έπρεπε να ασχοληθεί με τις διαφορές που παρατηρούνται στις διάφορες περιφέρειες και να ε, τις απαλείψει. Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες ε, ε, πλήγησαν πάρα πολύ και πρέπει λοιπόν οι γυναίκες αυτές να επανέλθουν στο προσκήνιο αυτών των ε, προγραμμάτων. Ε, για παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσω ε, της πρόσβασης, της ευκολότερης πρόσβασης σε πιστώσεις. Οι πολιτικές θα πρέπει να συνοδεύουν τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από την βρεφική μέχρι την τρίτη ηλικία. Ε, αυτά σε γενικές γραμμές. Ε, είχαμε καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση και τώρα και ύστερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, σκιώδης εισηγητής για τους ε, σοσιαλδημοκράτες δεν θα είναι η Βεραντάξ, δεν μπορούσε να ε, παραστεί στην σημερινή συνεδρίαση, όμως ε, μου έστειλε τις σημειώσεις της και θα τις διαβάσω. Η κυρία Ντάξ, λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστεί την κυρία Ντυπό για το εξαιρετικό της έργο όσον αφορά αυτήν τη γνωμοδότηση για τη ισότητα μεταξύ των δύο φίλων Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καλυφθεί και το κοινωνικό κενό και διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες. Πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε και στα δικαιώματα ΛΟΑΔΜ ΣΥΝ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία. Οι πρωτοβουλίε τώρα για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε διασυνοριακέ περιοχέ και σε ορεινέ περιοχέ είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό σύμφωνα με την έκθεση της Ρέγγι, αλλά δεν φτάνει. Υπάρχουν πολλές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου ε, λένε ότι δεν θέλουν να έχουν καθόλου ΛΟΑΔΜΟΥ. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε τέτοιες περιφέρειες με κοινοτικά κονδύλια. Η Επίτροπος Ντάλι απέρριψε έξι αιτήσει για χρηματοδότηση από διάφορες περιφέρειες ή πόλεις ή δήμους ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν επιπλέον από τα όσα τονίζετε κι εσείς στην γνωμοδότησή σας, κύριε Αντιπό. Οπότε, επιστρέφω στην ιδιότητά μου της Προέδρου και συνεχίζω δίνοντας το λόγο στην κυρία Σουζάνα Σόλης Πέρες από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντυπό για το έργο της όσον αφορά τη γνωμοδότηση αυτή. Πολύ χαίρομαι που συζητάμε στην Επιτροπή μας την έκθεση αυτή. Εγώ είμαι μέλος και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι πολύ σημαντικό τα κονδύλια συνοχής να χρησιμεύουν για πραγματικές αλλαγές σε διάφορες περιφέρειες. Τα αντιδροτικά ταμεία, είτε είναι το φεντερ, είτε είναι το κοινωνικό, αποτελούν το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και αποτελεί ένα πολύ βασικό εργαλείο επένδυσης για να βελτιωθεί η πολιτική μας όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Οι διάφοροι δείχτε δίνουν ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ακόμα και στο χώρο εργασίας και στο πολιτικό χώρο και στον κοινωνικό και οικονομικό. Οπότε η ισότητα αυτή πρέπει να είναι ένας εγκάρσιο στόχος. Όντω έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πετύχει πολλά, αλλά μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Από το Renew εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο υπέρ της ότας των δύο φύλων. Ότι οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ότας των δύο φύλων και να το λάβουν αυτό υπόψη τους σε όλο τον κύκλο της πολιτικής συνοχής από την προετοιμασία της μέχρι την υλοποίησή της και την χρηματοδότηση. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγές ε, των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών μελών και οι αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει συγκεκριμένων στόχων. Θέλουμε δεδομένα με ανάλυση για να μπορούμε να καταλήξουμε και εμείς σε συμπεράσματα για τις ανισορροπίες που υπάρχουν και να ξέρουμε ποια είναι τα προγράμματα εκείνα τα οποία λειτουργούν καλύτερα. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι η πολιτική συνοχή μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά τους προβλήματα όταν μιλάμε ιδιαίτερα για τις ε, περιφέρειες, τις ορινές, ή ε, εκείνες που έχουν μείνει με ελάχιστο κόσμο. Έτσι κι πρέπει να υπάρχουν παντού. η Γυροκομεία, φροντίδα για τα παιδιά. Μόνο έτσι θα βελτιώσουμε και την κατάσταση των γυναικών, οι οποίες πολύ συχνά αναλαμβάνουν και την φροντίδα των δικών τους έργο για το οποίο δεν αμείβονται έτσι κι αλλιώς. Και έτσι χειροτερεύει αυτό το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Χρειάζεται επίσης κατάρτιση, κάτι αναγκαίο για να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Κατάρτιση δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της συνοχής, ώστε να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ισότητας. Έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε η κρίση COVID-19 πόσο πολύ επηρέασε τις ζωές μας. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, για την οικονομία, για την υγεία και για την ισότητα. Και υπάρχει ένας κίνδυνος. Όσες χώρες επλήγησαν περισσότερο από την κρίση αυτή, θα έχουν λιγότερα χρήματα για να αγωνιστούν κατά των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να φροντίσουμε τα κονδύλια να πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται στις γυναίκες, στα παιδιά, με ισότητα απέναντι σε όλους. Νομίζω ότι η πολιτική συνοχή προφανώς αδιαφεσβήτητα μπορεί να βοηθήσει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη ισότητα των δύο φύλων σε όλου του τομεί εγκάρσια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ, Σουζάννα. Άννη πράσινη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Μόνικα Βάνα, αλλά και την Λένα Ντουπον για το έργο τους. Πραγματικά πρέπει να δούμε τώρα πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα οικονομικά μας εργαλεία υπέρ της ισότητας. Τώρα μάλιστα που ξέρουμε ότι με την πανδημία η ισότητα που προσπαθούμε να πετύχουμε πάει πίσω, γιατί με την πανδημία αυτή πάλι ένα μεγάλο βάρος πέφτει πάνω στις γυναίκες. Τώρα για την γνωμοδότησή σας κυρία Ντυπών. Συμφωνώ με πολλά από τα σημεία τα οποία συμπεριλαμβάνεται πρόθεση δηλαδή τις ισότητες μεταξύ των δύο φύλων, να μην υπάρχουν διακρίσεις από την πολιτική συνοχής, όντως και αυτό να ισχύει σε ολόκληρο τον κύκλο της πολιτικής συνοχής. Μ' αρέσει και αυτό. Στηρίζω και την ιδέα σας για να ενθαρρύνουμε συνεργασία ανάμεσα στην ε, ε, πολιτική συνοχής και το Ινστιτούτο για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι καλώ το Ινστιτούτο αυτό πράγματι, σωστά το είπατε και εσείς, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα δεδομένα που μας προσφέρει και πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε την πολιτική συνοχής. Μ' αρέσει και η πρότασή σας να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν την ισότητα των δύο φύλων όταν αναπτύσσουν τις πολιτικές τους σε περιφερειακό επίπεδο. Πολύ σωστό και αυτό. Και θέλω να στηρίσω και αυτά που πρότειναν οι συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές, δηλαδή να δούμε τι γίνεται με τις περιφέρειες αυτές, ε, δήμους πόλεις της Ευρώπης, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι περιοχές χωρίς ΛΟΑΔΜ, για παράδειγμα. Και να προτείνω και τρία πράγματα που ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ. Το ένα, να εκφράσουμε τη θλίψη μας που ισότητα μεταξύ των δύο φύλων δεν αναφέρεται σαν εκ των προτέρων όρος στον νεοκανονισμό. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθεθεί στην έκθεση ή τέλο πάντων είναι μια πρόταση που κάνω προς την εισηγήτρια. Δεύτερον, το πρόγραμμα γυναίκες σε ε, αγροτικές περιοχές στην Ήπεθρο. Η Επιτροπή ήθελε να το αποσύρει. Εμείς όχι. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και να αντικατοπτρίζεται αυτή η ιδέα στη γνωμοδότησή μας. Και τέλος, συμφωνώ απόλυτα με την τελευταία σας παράγραφο, η οποία έχει να κάνει και με αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τις γυναίκες την εποχή της πανδημίας, με προγράμματα, με ε, προσφορά φροντίδας, με κατάρτιση κτλ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη γνωμοδότηση. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ και πάλι για το έργο σας και ελπίζω και εγώ να έχουμε μια ιδιαίτερα ισχυρή γνωμοδότηση που θα βοηθήσει την εισηγήτρια της Επιτροπής επί της την κυρία Βάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κριστίν Άντερσον δεν έχει συνδεθεί, που είναι σκιώδης. ECR, Αγγέλικα Αναμοντανόφσκα. Δεν έχει συνδεθεί ούτε και εκείνη. Οπότε ευχαρίστως θα δώσω το λόγο στη Σάντρα Περέιρα που βρίσκεται στην αίθουσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και για μας είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα κονδύλια της συνοχής για να διαφυλάξουμε τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα κονδύλια και δημόσιες επενδύσεις για την καταπολέμηση της επισφαλείας και για να υπάρξει ε, εργασία με κάλυψη των δικαιωμάτων, ιδίω την προστασία της μητρότητας ή την ε, άδεια Επίσης, ο ίσος μισθός για ίδια δουλειά είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε, καθώς και να προωθήσουμε τις πολιτικές της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Θα πρέπει να δούμε ε, και το πλαίσιο της πανδημίας του COVID-2019 και να σκεφτούμε τι θα γίνει με την προστασία των αγροτησών, των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην γεωργία. Ιδίω με τις συνέπειες ε, του COVID-2019. Ε, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε ε, περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση της άμυνας και του στρατιωτικού εξοπλισμού και να περιορίζονται αυτά της παιδείας και της ε, κοινωνικής πολιτικής. Μας λείπουν τα χρήματα από την κοινωνική συνοχή, ενώ η στρατιωτικοποίηση και η διάσταση της ασφάλειας της κοινωνίας μας παίρνει όλο ένα και μεγαλύτερο βάρος εις βάρος των δικαιωμάτων των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σα Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 17 ε, Σεπτεμβρίου στι 5 το απόγευμα. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ο κύριος Μπιεντρών, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον, την εισηγήτρια για όλη τη δουλειά. Ε, την εκτιμούμε και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις για τα σχόλιά τους. Να σχολιάσω σύντομα όσα υπόθηκαν. Οι τοπικές κυβερνήσεις της Πολωνίας σε μερικές ε, περιοχές εγκρίνουν κάποιες εγκυκλίους και κάποιες αποφάσεις κατά τον ΛΟΑΚ και κατά της όπως έχει ονομαστεί ιδεολογίας τους. Αυτές οι περιφέρειες που εγκρίνουν τέτοια ψηφίσματα για αυτό που ονομάζουν ιδεολογία των ΛΟΑΚ δεν αφορά μόνο αυτή την ομάδα του πληθυσμού, εγκρίνουν και αποφάσεις που αφορούν τη διάσταση του φύλου. Δεν θέλουν τίποτε που να έχει σχέση με αυτήν την ε, αποκαλούμενη ιδεολογία. Αυτό καλό θα ήταν να αναφερθεί κάπου στο έγγραφο, διότι η θέση μας πρέπει να είναι ε, πραγματικά αυστηρή. Θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να προσφέρουμε ε, κονδύλια σε τοπικές κυβερνήσεις που υπονομεύουν τις πολιτικές της Ένωσης ακριβώς, ιδίως ως προς την ισότητα των φύλων. Αυτό που κάνουν αυτοί οι τοπικοί κυβερνήτες με τις κυβερνήσεις τους είναι να υπονομεύουν και να αμφισβητούν τη δουλειά μας. Έχουμε δυο λογιών λοιπόν αποφάσεις και κινήσεις από την πλευρά των κυβερνήσεων αυτών ε, κατά τον ΛΟΑΚ από τη μία και κατά της ε, ε, ισότητας των φίλων από την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο κάπως να φανεί συνεπές και να εγκρίνει μια συγκεκριμένη στάση και να ακολουθήσει πιστά μια γραμμή ως προς την κατάσταση αυτή. Ευχαριστούμε Ρόμπερτ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Παρόλο που έχουμε χρόνο μπορώ να το επαναλάβω βέβαια Θέλει η συγκητριά μας να ολοκληρώσει το γύρο αυτό των παρεμβάσεων. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τις ε, συνεισφορές σας και για τις πτυχές που θίξατε και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι επιθυμεί ο καθένα από τη δική του οπτική γωνία. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και να τα εντάξουμε στο ένα το άλλο σημείο θα σας ενημερώσουμε μαζί με την ομάδα μου για το πώς ακριβώς θα συνεχιστεί η μεταξύ μας συνεννόηση. Μάλιστα, η προθεσμία για την, ε, προθεσμία, η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι στις 29 Οκτωβρίου, αλλά θα επιβεβαιωθεί και αργότερα η ημερομηνία αυτή. Ε, ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης επίσης. Πάμε πολύ γοργά σήμερα και φτάνουμε κιόλας στο τέλος της συνεδρίασής μας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να ετοιμαστούμε για την συνεδρίαση των συντονιστών. Είστε έτοιμοι Ιδάλλως θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και να ξαναρχίσουμε. Ευχαριστώ όσους και όσες είσαστε εδώ στις Βρυξέλλες ή ήσασταν συνδεδεμένοι μέσω του, της πλατφόρμας Remote. Ευχαριστώ πολύ και τους διερμενείς και εμείς σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Ε, και θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για να κοιτάξουμε αν είμαστε έτοιμοι για τους συντονιστές. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ.